την έγκριση ενός πρακ, μιας πρακτικής λύσης για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίτροπε. Και γιατί ήσασταν λακωνικός. Και να περάσουμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Τομέα Αμήλου Γεωμήλων μετά το 2012. Για τρία λεπτά έχει το λόγο ως συντάκτρια της ερώτησης η κυρία Ντελάγκε. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, οι δύο ε, πιο μεγάλες ομάδες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΕΛΚ και η ομάδα των Σοσιαλιστών, ε, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν αυτή τη συζήτηση για το μέλλον του τομέα μήλου για ομήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μέλλον το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή λόγω και της χρηματοοικονομικής κρίσης και ε, ε, τίνει να εξαφανιστεί ο ε, κλάδος. Και ο κλάδος ακριβώς προσπάθησε να θέσει ε, κάποια ε, μέτρα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2020. Στα πλαίσια του Health Check ε, θα γίνει μερική αποσύνδεση ε, των ε, πληρωμών ε, και το 2012 θα έχουμε πλήρη αποσύνδεση. Mm. Πιστεύω ότι η παρούσα κατάσταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί καταλήλως για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να είναι ανταγωνιστικοί οι άλλοι κλάδοι. Ο κλάδος λοιπόν του τομέα του αμύλου γεωμήλων θα πρέπει να μπορεί να διεισδύσει στις αγορές, ε, κυρίως ε, στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων και θα πρέπει να είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να στοχεύσουμε στη στρατηγική μας. Θα πρέπει να σκεφτούμε ε, για παράδειγμα και τα πλαστικά τα οποία μπορεί να προκύψουν με βάση το άμυλο των γεωμήλων και να μην έχουμε μόνο πλαστικά από κατάλοιπα πετρελαιοειδών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε νέες αγορές και αυτό δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει, δεν υπάρχουν επενδύσεις για την καινοτομία και το 2012 δεν θα είναι γόνιμο το έδαφος ε, για τα θέματα αυτά. Ε, σύμφωνα με τις έρευνες θα χαθεί το 40% της αγοράς που κατέχει σήμερα και θα χαθούν και θέσεις εργασίας και άμεσες αλλά και έμεσες θέσεις εργασίας διότι θα πληχθεί ο τομέας εν γέννη και εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στην περιοχή μου εδώ αναφέρομαι και στη Δανία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Γαλλία Κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ένας συναγερμό, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να βοηθήσει τον κλάδο να πέσει στα μαλακά θα πρέπει να ληφθούν ε, μέτρα μέσως ε, για ένα διάστημα δύο ετών, ένα ε, μεταβατικό χρονικό διάστημα, το οποίο θα μπορέσει, για παράδειγμα, να σα επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε τις επιδοτήσει που δεν χρησιμοποιούνται στο γεωργικό τομέα και να προβλέψουμε και ένα ταμείο αναδιάρθρωσης για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς που θα ε, μειώσουν την παραγωγή τους επί εθελουσία βάσεω. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα το οποίο προκύπτει από αυτή τη συζήτηση. Θα θέλαμε ε, να ξέρουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σωστά λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο το άμυλο των γεωμήλων για τον τομέα της τεχνολογίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τον συνδράμουμε και να διασφαλίσουμε ότι θα περάσουμε στο μέλλον για τα θέματα στα οποία σας εξήγησα. Τώρα, για δύο λεπτά... Ο κύριος ε, Μπέρμαν. Να 2012 με έναν harde κλάπ in μια νέα περίοδο Κύριε Πρόεδρε, περνάμε από μια δύσκολη περίοδο και οι γεωργοί αυτοί θα περάσουν μια ακόμη πιο δύσκολα μετά το 2012 διότι πρόκειται για χίλιες θέσεις σε ένα ευάλωτο τομέα που δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λήξεις στο Γκρόνιγκεν και σε άλλες περιοχές πρόκειται για εργαζόμενους που δεν θέλουν να απομακρυνθούν από την περιφέρειά τους και θέλουν να συνεχίσουν να διαβιούν ε, στην περιοχή ε, όπου γεννήθηκαν ε, πράγμα το οποίο δεν θα κοστίσει διότι υπάρχουν ακόμη υπολείμματα από τις επιδοτήσεις τις περισσινές και τις προπέρσινες και θα επιτρέψουν στους ε, ε, γεωργούς να ε, προσαρμοστούν. Βέβαια το 2012 θα εξαφανιστούν οι επιδοτήσεις για το άμυλο γεωμήλων αλλά εντωμεταξύ θα πρέπει να δώσουμε εναλλακτικέ ρήξει για διαφορετικά προϊόντα όπως το λάδι που θα επιτρέψουν σε αυτούς τους γεωργούς να επιβιώσουν. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπέρμαν. Ο Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις για το μέλλον του τομέα μήλου ομήλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται που μπορεί να εκφράσει και αυτή την άποψή τη επί του θέματος. Ο τομέα αυτό ήταν τμήμα του Health Check και είχε ζητηθεί από τον τομέα ε, να αποφασίσει για την αποσύνδεση των πληρωμών και αποφασίστηκε όντως αυτή η αποσύνδεση ταυτόχρονα με την κατάρρευση του συστήματος των ποσοστώσεων. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόβλεψε αποσύνδεση σε δύο στάδια. Τα επιχειρήματα του τομέα ήταν ότι επιπλέον καθυστέρηση ε, θα επιτρέψει να έχουμε μία αγορά χωρίς ε, ποσοστώσεις και χωρίς ε, επιδοτήσεις για αλλαγή εκμετάλλευσης και αυτό το μεταβατικό στάδιο θα ήταν πιο ομαλό. Ακόμα και αν όλοι ασχολούνται με τον τομέα του αμήλου των γεωμήλων αποφασίσουν να μην λάβουν τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή για να συσταθεί ένα ταμείο αναδιάρθρωσης, ο προ βλεπόμενος προπολογισμό κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αρκεί. Τα... Ε, οι επιδοτήσεις ε, βέσω των διαστατικών ταμείων προβλέπουν ένα συγκεκριμένο κανονισμό ο οποίος δεν μπορεί να υπάρξει πριν από το τέλος του 2011 που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα ταμείο αναδιόρθωσης με πολύ περιορισμένο προπολογισμό που δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που βάσει του τομέα μπορεί να φτάσουν μέχρι και στο 40% της παραγωγικότητας που έχουν αυτή τη στιγμή. Όπως ανέφερα πριν, νωρίτερα για την απόφαση η οποία λήφθη από το Health Check δεν ε, πρόκειται για εναλλακτική λύση. Εξετάζουμε τι μπορεί να γίνει μετά το 2013 και για τον τομέα της γεωργίας θέλουμε να έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική που θα είναι αποτελεσματική και ισορροπημένη. Και φυσικά το θέμα του αμήλου γεωμήλων μπορεί να συμπεριληφθεί σε όλη αυτή τη συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε τον Επίτροπο, να περάσουμε τώρα στις πολιτικές ομάδες, εξ ονόματος του ΕΛΚ για τρία λεπτά ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Με ε, τον ε, κανονισμό αυτό για τις ε, άμεσες πληρωμές για τη γεωργική πολιτική άλλαξαν, η, άλλαξε το σύστημα και αποδεσμεύτηκαν οι πληρωμές ε, υπάρχουν όμως ακόμη ορισμένα στοιχεία που μπορούν ε, να ε, χρησιμοποιηθούν σαν συνδεδεμένες πληρωμές για την πληρωμή των γεωργών και των εργοστασίων θα μπορούσαν λοιπόν να αποσυνδεθούν αυτές οι πληρωμές και να χρησιμοποιηθούν οι ενισχύσεις αυτές. Πράγμα το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει σε μία αποσύνδεση από το 2010. Πράγμα το οποίο θα επιτρέψει ε, το άμυλο γεωμήλων να συνεχίσει να παράγεται αλλά μετά από τον έλεγχο υγείας έχει διαπιστωθεί ότι θα πρέπει η παραγωγή αυτή να ανασταλεί καλεί το αργότερο το 2012 ε, το εάν η ε, η καλλιέργεια αυτού του αμύλου για έχει μέλλον ή όχι είναι κάτι που θα πρέπει να ερευνηθεί πρέπει να δούμε αν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις και να εξευρεθούν μεταβατικές περίοδοι για να υπάρξει μία προσαρμογή γι' αυτό και οι γεωργοί οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν πρέπει να βοηθηθούν να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους και να διερευνήσουν εναλλακτικέ αγορές αλλά ε, το πιο βασικό από όλα αυτά είναι βραχυπρόθεσμα να γίνει μία σαφής δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση. Μία καλή απόφαση είναι πάντοτε καλή, η κακή είναι πρόκληση, αλλά καμία απάντηση και απόφαση ε, ε, είναι στασιμότητα που σκοτώνει την γεωργία. Παρακαλώ λοιπόν Λοιπόν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα το ταχύτερο δυνατόν για να βοηθηθούν οι γεωργοί μας. Ευχαριστούμε κύριε Γιάρ. Για τους φιλελευθέρους, για 1,5 λεπτό, ο κύριος Μούλτερ. Κύριε Πρόεδρε, σε έναν ιδεώδη κόσμο, για να το πω έτσι, δεν θα υπήρχαν τα προβλήματα που συναντάμε στον τομέα του αμήλου των γεωμήλων. Διότι εκεί απειλούνται με πτώχευση πολλές εταιρείε λόγω της χαμηλοτάτης τιμής του γεωμήλου. Αυτό είναι το πρόβλημα, η τιμή. Η τιμή. Έχουν γίνει και ορισμένες πρόοδοι βιοχημικός. Δημιουργήθηκαν νέα προϊόντα και αυτή η πρόοδος δεν πρέπει να εμποδιστεί. Οι προτάσεις της Κομισιόν δεν μας επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία. Ερωτώ λοιπόν, θα επανεκτιμήσετε τα πράγματα, Ο, θα κάνετε διάλογο με τους προσώπους του τομέα, διότι νομίζω ότι για να μπορέσουν οι γεωργοί να έχουν κάποια λύση χρειάζεται επαναδιαπραγμάτευση. Το άμυλο του γεωμήλου είναι κάτι το τελείως ιδιαίτερο και πρέπει να μπορέσει να επιβιώσει. Άρα να πάρετε όλος εξαιρετικά μέτρα και για αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε κύριε Μούλντερ, ο κύριος και για την ομάδα του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά την προηγούμενη θητεία δύο φορές ήμουν εισηγητής για το πρόβλημα των ποσοστώσεων του αμήλου γεωμήλων και γι' αυτό είχα συνεννοηθεί με προσώπους του τομέα και προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τις ευχές τους που διαφωνούσαν βέβαια με τις ποσοστώσεις που είχαν καθοριστεί και γι' αυτό έπρεπε να βρεθεί μια άλλη ισορροπία. Αυτή τη στιγμή ακούμε ότι απειλείται πάλι ο τομέας και ότι μπορεί και να εξαφανιστεί τελείως. Αυτό με λυπεί ιδιαίτερος. Διότι εδώ βλέπουμε ότι τομέα με τον τομέα τα ίδια γίνονται και στο γαλακτοκομικό, τα ίδια στη ζάχαρη, στον καπινό και τώρα στο άμυλο του γεωμήλου. Όλοι οι τομείς το ίδιο πρόβλημα λοιπόν έχουν και πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα σφαιρικά. Ίσως να χρειαστούν νέες κατευθυντήριες γραμμές, ίσως οι βασικές αρχές δεν μην ισχύουν πια. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η οφθαλμοθυρία. Ο κύριος Καλινόφσκι για ένα λεπτό. Στο πολύ κύριε Πρόεδρε. την περιοχή μου άμυλο γεωμήλων παράγουμε εδώ και πολλά χρόνια και όπως και άλλοι παραγωγείς φοβόμαστε και εμείς ότι άμα αποσυρθούν οι επιχορηγήσεις στην παραγωγή αυτή και στη μεταποίηση θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα και τεράστια προβλήματα. Το 2013 νομίζω ότι η κατάσταση θα καταστεί κρίσιμη. Θα ήθελα λοιπόν να διατηρηθούν τα υπάρχοντα εργαλεία στήριξης του αμήλου γεωμήλου. Γιατί πρέπει να υπάρξει μία τουλάχιστον ελάχιστη στήριξη των τιμών. Αφού και για τη ζάχαρη κάναμε συγκρίσεις πρέπει να πω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύουν τα ίδια για το άμυλο. Η μεταρρύθμιση του τομέα ζάχαρης ήταν τρομερή αποτυχία. Ευχαριστούμε κύριε Καλινόσκη. Τώρα για ένα λεπτό πάλι κυρία Κούστινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 20% λιγότερα ε, διοξίδιο του άνθρακος και ε, ε, μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτά επιζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να έχει εξοικονόμηση ενεργείας. Αλλά πώς θα γίνουν αυτά. Η γεωργία δεν μπορεί να ε, μην συμβάλλει τη βασική της συμμετοχή στους στόχους του 2020. Ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν ε, να δημιουργεί κανείς κατά τον έλεγχο υγείας της γεωργίας συνθήκες ή στον τομέα του αμύλου γεωμήλων όπου δημιουργούνται φοβερές πιέσεις για τους γεωργούς πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλιστεί η παραγωγή του αμύλου γεωργίων για ορισμένες περιοχές που εξαρτώνται από αυτό διότι θα έχει σημαντική σημασία αυτή η παραγωγή για το μέλλον. Κύριε Κέλλη, ε, είναι η τρίτη φορά που ε, πιάσατε το, το, την προσοχή μου. Ε, ξέρετε τι λένε. Λένε ότι όποιος ξυπνάει νωρίς βγαίνει κερδισμένος. Το βράδυ όμως μπορούμε να προσελκύσουμε την προσοχή του Προέδρου. Και πρέπει να πω ότι το 1947 πέθαναν 4.000 άτομα όπου δεν είχαμε καλή εσοδεία πατάτα στην Ιρλανδία. Έκτοτε λοιπόν πρέπει πάντοτε να υπολογίζουμε την πατάτα και γι' αυτό τα τελευταία μέτρα μας έκαναν να ανατριχιάσουμε. Ε, ανησυχούμε πάρα πολύ για το μέλλον της βιομηχανίας της πατάτας διότι λέγεται ότι μετά το 2013 η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να αναθεωρηθεί ε, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι σας ε, συγχαίρω ε, για την προεδρία σας απόψεις και αν δεν ήμουν αντίθετος προς την κλωνοποίηση θα ζητούσα να κλωνοποιηθείτε εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο Επίτροπος τώρα. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συμφωνώ με την άποψή σας ότι ο τομέας του αμύλου και ομίλων μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για την παραγωγή βιοπλαστικών και άλλων ε, συναφών προϊόντων. Βιοπλαστικών. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και το ε, πλαίσιο προπολογισμού και το νομοθετικό πλαίσιο και φυσικά το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να συνδράμουμε τον τομέα. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας θα λάβει μια μελέτη για τα γεώμηλα και το άμυλο των γεωμήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη και τη συζήτηση για την ε, μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής μετά το 2013. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να βρούμε μια πιο βιώσιμη και πιο σταθερή λύση και ε, από τα ε, στοιχεία που έχουμε βάσει του τρέχοντος πλαισίου. Κύριε Λάγκε, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν ήσασταν στον κατάλογο. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πολύ σημαντικό, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να πω στον κύριο Κέλλη για τα όσα είπε για τα γεώμελα. Εμείς μιλάμε για άλλο είδος γεωμέλων. μιλάμε για το άμυλο των γεωμήλων. Είναι όμως αλήθεια ότι τα προβλήματα είναι αλληλένδετα. Ο τομέας ε, του αμύλου των γεωμέλων καταραίει. Και αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις ε, και στην παραγωγή και στην κατανάλωση πατάτες και είναι αλήθεια ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Θα πρέπει όμως να εξεύρουμε μία λύση ας προσπαθήσουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Ο Επίτροπος όταν αναφέρεται στο διάστημα μετά το 2012, για το 2013 δηλαδή, ε, χρονοτριβή. Πρέπει να παρέμβουμε αμέσως, διότι ο κίνδυνο είναι άμεσο και μπορεί να καταρρεύσει ο κλάδος του αμήλου και ομήλων ε, Ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε λάβει κάποια μέτρα για να είμαστε σε θέση να συζητήσουμε το 2013. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Έχετε δικαίωμα να κλείσετε εσείς τη συζήτηση. Όχι. Ωραία λοιπόν. Πολύ καλά. Εξαντλήσαμε και το θέμα αυτό.